Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten noch einige. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν απόλυτα στην ώρα μου. Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση για τα θύματα της τρομοκρατίας στη Βόρεια Ιρλανδία. Αγαπητοί συνάδελφοι,